Καλή σας μέρα. Ακολουθεί ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τη διανομή τροφίμων στα πλέον άπορα άτομα της Ένωσης. Το λόγο έχει ο Επίτροπος, κύριο Σολιρέν. Uh, Πρόεδρε. Σημειώνω